Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Άρχεται η συνεδρίαση. Συνεχίζεται η συνεδρίαση μετά την διακοπή 25 Νοεμβρίου του 2010. Έχετε το σχέδιο των πρακτικών. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, εγκρίνονται. Θα ήθελα να κάνω κάποιες προκατακτικές ανακοινώσεις πριν περάσουμε σε εργασίες μας. Η διάσκεψη των Προέδρων την περασμένη Πέμπτη έλαβε κάποιες αποφάσεις. Αύριο στις 4 η ώρα θα κάνουμε μία συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Ιδονία Ζενιέσκα και της κυρίας Τρίπελ για το νέο σχέδιο προϋπολογισμού του 2011. Έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία για την Τετάρτη. Δεύτερη ανακοίνωση, αύριο θα γίνει συζήτηση για τα αποτελέσματα της COP16, της διάσκεψης της Κανκούν για τις κλιματικές αλλαγές. Σημειώθηκε πρόοδος στην Κανκούν και ένα κλιμάκιο του Κοινοβουλίου φυσικά συμμετείχε στη διάσκεψη. Οι συνάδελφοι είναι σήμερα μαζί μας και από κοινού με την Επίτροπο θα συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε τελικά να αποβεί επωφελής η συμφωνία ε, και θα προετοιμάσουμε τη διάσκεψη στη Νότιο Αφρική. Ε, στις 21 Οκτωβρίου μάθαμε για το βραβείο Ζαχαρόφ, για την ελευθερία της σκέψης. Ο Γκυγέρμο Φαρίνιας κέρδισε το βραβείο Ζαχαρόφ. Δυστυχώς ο κύριος Φαρίνιας κολλείεται ε, για να μεταβεί στο Κοινοβούλιο και να παραλάβει αυτοπροσώπως ε, το βραβείο. Επέμεινα εγώ ίδιος ε, και έστειλα επιστολή στον κύριο Ραούλ Κάστρο. Προς το παρόν είναι αδύνατο να γίνει κάτι και λόγω του ότι ο κύριος Φαρίνιας δεν μπορεί να μεταβεί στο Κοινοβούλιο, υποθέτω ότι η κυρία Άστον θα λάβει υπόψη την κατάσταση δοθέντων και των σχέσεων που έχουμε με την Κούβα. Ευελπιστούμε ε, ότι θα μπορέσει τελικά να έρθει εάν φύγει τις προσεχείς ώρες ε, από την Κούβα θα μπορούσε να φτάσει εγκαίρος ε, για την απονομή. Κατόπιν στις 13 Δεκεμβρίου 81, πριν 20 χρόνια, κηρύχθη η πολιορκία στην Πολωνία και προσπάθησε η κομμουνιστική κυβέρνηση ε, να ε, επιδείξει αλληλεγγύη ε, Είχαμε πάνω από 100 θανάτους, πολλούς τραυματίες. Πέρασαν όλες αυτές οι δεκαετίες ε, και αποτείουμε φόρο τιμής για όσους αγωνίστηκαν για να ελευθερώσουν την Ευρώπη. Πέμπτη ανακοίνωση. Ε, δοθεί η συμπεριφορά του κυρίου Μπλουμ στην τελευταία ε, σύνοδο Ολομέλειας και λόγω του ότι βάσει του άρθρου 9 και 153 του κανονισμού ε, δεν απολογήθηκε, ε, άρα αποφασίζω ότι για 7 ημέρες δεν θα λάβει την ημερήσια αποζημίωση στο diem. Έχω ενημερώσει ε, προσωπικά και τον κύριο Μπλουμ για αυτή μου την απόφαση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να σας ενημερώσω για την υπογραφή πράξεων βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Την Τετάρτη ο Πρόεδρος Συμβουλίου και εγώ θα υπογράψουμε μια δεκάδα τέτοιες νομικές πράξεις ε, βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 74 του ιστορικού κανονισμού και θα δημοσιευθούν αυτές οι νομικές πράξεις στα πρακτικά της παρούσας ε, συνόδου. Κατόπιν η κυρία Πάσκαλ Γκρινή με ενημέρωσε γραπτός ε, ότι εκπνέει η θητεία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι εξελέγει στην Γαλλική Βουλή. Βάσει του άρθρου λοιπόν 7 παράγραφος 2 όπου ε, προβλέπονται διατάξεις περί εκλογών και βάσει το άρθρου 4, παράγραφος 1 και 4 του κανονισμού, του ιστορικού κανονισμού, αποφασίζουμε ότι χειρεύει πλέον η έδρα της από 14 Δεκεμβρίου 2010 και μετά κατόπιν. Η ομάδα ε, των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων μου ζήτησαν ε, να διορίσω τον κύριο Γιωχάνης Κορνέλης Φανμπάλεν στην διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν θα αντικαταστήσει τον κύριο Καρλ Χάγκλουντ. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Οπότε εγκρίνεται ο διορισμός του. Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη τώρα. Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξη που έγινε δεκτό από την διάσκεψη των Προέδρων στις 9 Δεκεμβρίου δυνάμει του άρθρου 137 του εσωτερικού κανονισμού δημοσιεύτηκε για τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν υπάρχει καμία αλλαγή, καμία εισήγηση, καμία... οπότε θα περάσω κατευθείαν στην Τετάρτη. Η ομάδα ΕΛΚ ζήτησε την προσθήκη του κυρίου Σάγερ για τον έλεγχο που διεξάγουν τα κράτη-μέλη ως προς την άσκηση κάποιων αρμοδιοτήτων, εφαρμοστικών ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Σάγερ, σας δίνω το λόγο. Πρόεδρε, όπως είπατε σωστά, ζητούμε να μπει στην ημερήσια διάταξη ο κανονισμός για την εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων της Επιτροπής και είναι κάπως παράξενο αυτό. Δεν είναι αίτημα μόνο τη ομάδα μου. Και άλλες ομάδες υποστηρίζουν την ιδέα αυτή. Και στην νομική επιτροπή